Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Βάσει της ημερησίας διάταξης προχωρούμε στην κοινή συζήτηση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Καταστατικό της Ρώμης. Με την έκθεση του κύριου Ραμών Χαουρέγγι, για τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την διάσκεψη για την αναθεώρηση του καταστατικού της Ρώμης σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Καμπάλα της Ουγκάντα. Δίδω αμέσως το λόγο στον εισηγητή κύριο Χαουρέγγι για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Νομίζω ότι η μέρα αυτή είναι μια σημαντική μέρα. Ξέρω ότι πολλές είναι